So, dear colleagues, maybe we could continue. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρτε θέσει για να ξεκινήσουμε. Θέλω να επανέλθω στο πρώτο σημείο τη μέσης διάταξη τη αποφάση των συντονιστών. Σήμερα το πρωί οι συντονιστέ πήραν τι εξή αποφάσει να ορίσουν τον κύριο Καβαντά ως εισηγητή μετά το αίτημα ενός waiver για να αρθεί η ασυλία της κυρίας Μόνικα Χοκμάιερ να εγκρίνουμε τις συνειδριάσεις ε, από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο του 2019 και με βάση το, το κανόνα 39 παράγραφος 3 να εξεταστεί κατά πόσο είναι σκόπιμη η προτινόμενη νομική βάση άρθρο 53 παράγραφος 1 και άρθρο 62 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη προσωρινή συμφωνία σχετικά με, με το φάκελο ΣΑΤΚΑΜ. Τώρα, κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Συνεδρίου για την εισφορά στο πρόγραμμα εργασιών του, του, 2020, ε, πάρθηκε και αυτή η απόφαση και πάρθηκε η απόφαση να καλέσουμε και τον, τον Επίτροπο Άνσιπ τον Φεβρουάριο, αντί να οργανώσουμε ακρόαση για την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω δύο κρατών διαδικασιών στην τρίτη εβδομάδα οι συντονιστέ αποφάσισαν να συμφωνήσουν ότι θα σταλεί μια ε, επιστολή για, με τη γνώμη μας για τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργίας και να ακολουθεί μια προστατευμένη διαδικασία του άρθρου 50 παράγραφος 1 των, του ιστορικού κανονισμού και να οριστεί, να οριστεί ο κύριος Βιέρκα ως εισηγητής για την, την επανεξέταση του Recast Βρυξέτες 2α. Αυτά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών. Μπορούμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με το σημείο 6 ανταλλαγή απόψεων ακριβώς για την αναδιατύπωση του Βρυξέλλες 2α. Recast. Και βεβαίως έχουμε εδώ την επαναδιαβούλευση. Κύριε Ζιεύκα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, poinformował rzeczywiście mm, Όπως είπε ο Πρόεδρος temat rozporządzenia Bruksela 2 mm, Στην Βρυξέλλες 2α είχαμε κάποιες περαιτέρω συζητήσεις έχουμε φτάσει τώρα στην επαναδιαβούλευση το Συμβούλιο απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτό το αίτημα να λάβουν χώρα δηλαδή, διαβούλευσης ε, για το συγκεκριμένο έγγραφο. Το έγγραφο όμως αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. σε ό,τι αφορά τα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εδώ και δύο χρόνια εξετάζει το ζήτημα και έχει αλλάξει σημαντικά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την έχει τροποποιήσει. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ ζητείται από το Κοινοβούλιο ε, μια διαβούλευση εκ νέου, έχει ξαναγίνει αυτό το παρελθόν. Τι συμβαίνει όμως, έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Βεβαίως ε, θα είχατε την ευκαιρία να δείτε ε, πόσο οι συντονιστές ε, ε, μου ανέθεσαν να αναλάβω την επόμενη έκθεση την προετοιμάζω ο κύριος Βόμποντα ο πρόεδρος και εφόσον η προθεσμία που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ μικρή μέχρι να τελειώσει δηλαδή η θητεία μας πρότεινε το εξής ο πρόεδρος να ακολουθήσουμε το άρθρο 50 ε, του εσωτερικού κανονισμού, αυτήν δηλαδή την ε, γρήγορη διαδικασία, ε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κυρίε και κύριοι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε άμεσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα δεν θα υπάρξει πολλής χρόνος για ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει γρήγορα να εγκριθεί αυτή η έκθεση. Θα είναι σύντομη αυτή η έκθεση. Τι θα σας την παρουσιάσω. Αν μου το επιτρέπετε, θέλω να αναφερθώ πρώτα στις εργασίες του Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κάναμε και εμείς ως Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Εμείς έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερα ζητήματα θα έλεγα. Πρώτον, η διαδικασία της εξεκουάτου ε, θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι είναι τεχνικό το θέμα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Διότι αυτός ο κανονισμός ρυθμίζει μια σειρά από εξαιρετικά λεπτά ζητήματα. Τώρα τα πλέον σημαντικά θέματα στον κανονισμό. Εμείς βασιστήκαμε στις συζητήσεις με τους εμπειρογνώμονες και εδώ Είχαμε συζητήσει και με του εκπρόσωπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και είδαμε ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι πρέπει είναι πολύ σημαντική η γνώμη του παιδιού, να ακουστεί η γνώμη του παιδιού, να, να υπάρξει διαδικασία τη διαμεσολάβησης και στις διαδικασίες όπου υπάρχει ε, αντιπαράθεση στο ιστορικό της οικογένειας ε, όπου υπάρχει δηλαδή διένεξη, θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Βεβαίω υπάρχουν και τα ζητήματα τις περιπτώσεις, οι περιπτώσεις εκείνες όπου το παιδί δεν είναι με την οικογένειά του ότου πάρθει μία απόφαση. Εμείς πάντα έχουμε κατά νου πρωτίστως το καλό του παιδιού. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να βρίσκεται κάθε φορά η καλύτερη λύση για το πιο εύθραυστο, το πιο αδύναμο κρίκο σε αυτή την αλυσίδα, το παιδί δηλαδή. Αυτό ήταν πάντα στο κέντρο των ανησυχιών μας και για όλα αυτά τα ζητήματα το Συμβούλιο έχει δεχθεί αυτή την ιδέα που τους είχαμε, που τους είχαμε υποβάλει. Το Συμβούλιο έχει φέρει ένα νέο άρθρο σχετικά με τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Και εδώ ε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Τι έκανε το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προσπάθησε να περιγράψει μια σειρά από περιπτώσεις που προκύπτουν στην πραγματικότητα. Ξέρετε ότι ως νομοθέτες ε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα κανόνα για την κάθε περίπτωση, αλλά μπορούμε να ομαδοποιήσουμε ε, κάποιες περιπτώσεις. σε ένα νομοθετικό έγγραφο. Αυτό βοηθάει στο να βελτιωθεί το έγγραφο αυτό. Το Συμβούλιο λοιπόν αφιέρωσε πολύ χρόνο ξέρετε το στο Συμβούλιο ε, με τα κράτη-μέλη αυτό παίρνει χρόνο ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ζητήματα γενικού δικαίου, ε, είναι δύσκολο. Ιδιαίτερα πρέπει να βρεθεί μια διασυνοριακή λύση ε, Εν πάση περιπτώσει κατέληξε το Συμβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κείμενο είναι ολοκληρωμένο, έχει ολοκληρωθεί, έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα, τα θεσμικά όργανα, βελτιώνεται έτσι η κατάσταση σε νομικό επίπεδο και η νομική σαφήνεια, η νομική ασφάλεια τον τομέα αυτό. Μιλάμε για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών εδώ, δημιουργούνται κάποια νομικά μέσα ε, σε επίπεδο κρατών μελών ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις που θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες από τη μία χώρα στην άλλη σε ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση την οποία σας υποβάλλω. Πρέπει να πω ότι εμείς ως Ευρωπαϊκοί ε, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή τη δουλειά. Επειδή λοιπόν ακολουθείται η γρήγορη διαδικασία έτσι ώστε να εγκριθούν όλα αυτά πριν την ολοκλήρωση της θητείας μας, να κάνουμε αυτές τις αλλαγές τις οποίες αναφέρθηκα ε, στον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, η έκθεση που σας υποβάλλω κυρίες και κύριοι είναι εξαιρετικά σύντομη. Τι λέμε εδώ. Ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται επί της ουσίας, την πρόταση του Συμβουλίου. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι στη συνεδρίαση αυτή θα γίνει μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας εδώ. Εάν θέλουμε να εγγυηθούμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε βήμα-βήμα Πιστεύω ότι στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση, μια μικρή συζήτηση για το θέμα αυτό που θα περιοριστεί σε ένα γύρο παρεμβάσεων από τις πολιτικές ομάδες ε, και ως εκεί. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έτσι θα έχουμε και λίγο χρόνο να ακούσουμε ε, τις απόψεις των πολιτικών ομάδων αλλά να σεβαστούμε ταυτόχρονα και το χρονοδιάγραμμα. Η διάσκεψη των Προέδρων θα μπορούσε να πάρει αυτή την απόφαση και να προχωρήσουμε. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίω ε, κύριε Πρόεδρε είμαι στη διάθεσή σας ε, για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την γρήγορη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκέμπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και τον κύριο Τσβιεύσκα που ε, είχε ε, ήδη από την αρχή φροντίσει να συμμετέχουμε εμείς ε, οι συγγητές ε, και μας διαβουλεύτηκε από την αρχή και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερος. Πραγματικά είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι το Συμβούλιο για μια ακόμη φορά ξεκινά διαβούλευση. Δεν ήθιστε να το κάνει και ξέρετε ότι το έχουμε ζητήσει από το ψηφισμά μας και έχουμε ζητήσει να γίνεται αυτό εάν προβεί το Συμβούλιο σε αποφασιστικές αλλαγές προτάσεις της Κομισιόν. Άρα αυτό είναι κάτι θετικό. Και αυτό αυτή η νέα ρύθμιση Βρυξέλλης 2α είναι κάτι πολύ σημαντικό, ε, είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα και συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή ότι δηλαδή ε, πρέπει να ακολουθήσουμε μια ταχεία διαδικασία ώστε στο πλαίσιο της τρέχουσας θητείας να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθετική διαδικασία, διότι πρόκειται για την ευμερία των παιδιών σε περίπτωση που έχουμε διεθνείς ε, ε, αρπαγίες παιδιών ε, και θα πρέπει να δούμε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, αν μπορούμε να λύσουμε με εύλογο τρόπο τα προβλήματα αυτά και επομένως νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ταχεία διαδικασία. Είναι λοιπόν ένα θέμα σημαντικό και σίγουρα πρέπει να γίνει συζήτηση ε, στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Γι' αυτό συμφωνώ και με αυτή τη ε, διαδικασία που μόλις μας πρότεινε ο εισηγητής, ε, δηλαδή αναπολιτική ομάδα να έχουμε έναν καλεσμένο και να γίνει μια ανταλλαγή απόψε ένας γύρος ή μάλλον ένα άτομο από κάθε πολιτική ομάδα να μιλήσει ώστε να γνωρίζουμε περισσότερα. Ε, σε ό,τι τώρα αφορά το περιεχόμενο, τρία σημεία ε, είναι αυτά τα οποία θα ήθελα πιο πολύ να σχολιάσω, αυτά τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα ανέφερε και ο εισηγητή μα, ο κ. Σβιεύσκα. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχω διατελέσει και διαμεσολαβήτρια για τις διασυνοριακές ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις, έχω ε, ε, για το άρθρο 23α. Ε, τι γίνεται σε περίπτωση ε, που το συσχετίσουμε με τις αρπαγές παιδιών. Έχουμε ένα άλλο μοντέλο προτείνει ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν συνάδει με την πρόταση αυτή και πιστεύω ότι όλοι οι γονείς θα έπρεπε ακριβώς λόγω του καλού του παιδιού τους ε, να κάνουν ένα διάλογο για να καταλήξουν ε, σε αυτό που θα ήταν καλύτερο στην κάθε περίπτωση για το παιδί. Και καλό θα ήταν ε, να υπάρχει επαφή του παιδιού και με τους δύο γονείς. Ιδίως βέβαια αν δεν υπάρχουν περιπτώσεις ε, βίας και κακοποίησης του, του, παιδιού. Αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει επαφή το παιδί και με τους δύο του γονείς για να ε, μπορούν και οι δύο να τα τρέφουν. Επίσης έχουμε ε, το 1 α που αλλάζει τον ορισμό το Συμβούλιο και ε, δεν αφήνει τη λήψη αποφάσεων στις αρχές. Ε, αλλά στα δικαστήρια που σίγουρα είναι, έχουν τη νομική δικαιοδοσία για να λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά θεωρώ ε, και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό. Και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες ε, για την περίπτωση της γονικής ευθύνης και κάποιες αποφάσεις, όλα αυτά τα οποία γράφει το Συμβούλιο σε αλλαγές ε, της τροποποίησης, νομίζω ότι ε, είναι πολύ πιο διεξοδικά σε σχέση με τα όσα είχαμε προτείνει εμείς ως Κοινοβούλιο, αλλά φαίνουμε, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η εγκύτητα με το τι ισχύει στην πράξη, ε, πολύ περισσότερο από ό,τι πριν και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και πρέπει να πω ότι είναι και καλύτερο από αυτό το οποίο είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο προτείνει δηλαδή τώρα το Συμβούλιο. Για να ληφθούν υπόψη ναι, ε, τα διαφορετικά δεδομένα και αυτό το θεωρώ πολύ θετικό. Και το εξεκβάτουρ, ε, το τέταρτο σημείο, δεν θα το σχολιάσω γιατί το είπατε και εσείς, το καλύψατε παρκώς. Τώρα, καταλήγω Γοντάς θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω με τη διαδικασία αυτή. Δεν θα καταθέσω εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας καμία τροπολογία για να μην τεθεί σε κίνδυνο η όλη διαδικασία και προκειμένου να προχωρήσουμε με την ταχεία διαδικασία, όπως ε, είπα και πριν. Απλά υπάρχουν κάποια σημεία που λείπουν και για μένα και την δική μου πολιτική ομάδα έχουν σημασία. Έχω λοιπόν κάποια ερωτήματα και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς το Συμβούλιο. Και αυτά τα ερωτήματα θα τα θέσω. Πρέπει να πω ότι ζούμε σε μια σύγχρονη κοινωνία και γι' αυτό το λόγο διαρωτώ. Γιατί μόνο για ένα ε, τμήμα του πληθυσμού έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις στο 2α, ε, Βρυξέλλες 2α, γιατί μόνο για τους ε, ε γάμους ναι, ισχύει και όχι για τα σύμφωνα συμβίωσης, ε, εφόσον αλλάζουν τα πράγματα στην κοινωνία. Θα ήθελα να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μου απαντήσει και το Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό. Και μια άλλη ερώτηση που έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες 2α. Ε, υπάρχει στο προβλέψο μέλλον κάποια ε, πρόθεση επέκτασης του πεδίου ο εφαρμογής για να μην καλυπτονται μόνο τα ζευγάρια που έχουν συνάψει γάμο, γιατί αυτό στα διακριτική μεταχείριση μεταξύ των ζευγαριών. Το ε, ε, ερώτημα απευθύνεται και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, ώστε λοιπόν στα σύμφωνα ε, συμβίωσης να υπάρξει αυτή η επέκταση να καλύπτονται, έστω αν συζητείτε καν αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Επίσης, το Βρυξέλλες ΔΑ θα ήθελα να έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει τα ελάχιστα πρότυπα και για τις ακροάσεις των παιδιών. Το είχαμε προτείνει, δεν το έλαβε υπόψη το Συμβουλίο τελικά. Όπως είπα όμως έχω διατελέσει ε, διαμεσολαβήτρια κατά τον παρελθόν εκ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου η ακρόαση ενός ε, παιδιού πήγε ε, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ήταν μια τραυματική εμπειρία για το παιδιό. Γι' αυτό θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μεταλάβουμε να καταλήξουμε σε κάποια ελάχιστα πρότυπα για τις ακουράσεις των παιδιών και τα κράτη-μέλη νομίζω ότι θα πρέπει να ε, το λάβουν αυτό υπόψη στο και των αρμοδιοτήτων της Επομένως, ό,τι αφορά τη θέσπιση κατώτατων του προτύπων για την ακρόαση, υπάρχει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή στην Κομισιόν ή λείπει η πολιτική βούληση επ' αυτού. Θα ήθελα και θα μπορούσα ε, και θα το έκανα με μεγάλη χαρά να καταθέσω πολλές τροπολογίες, αλλά όπως σας είπα, επειδή πλησιάζει το τέλος τέλος της θητείας και δεν θα ήθελα να θέσω σε κίνδυνο τα όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αντίθετα να τα διασφαλίσω. Ε, αν είμαι στην επόμενη θητεία εδώ, θα παραμείνω σε επάλξεις και θα φροντίσω το θέμα αυτό να ξανασυζητηθεί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα ήθελα μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλες και όλους. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την πρώτη νομοδότηση του Κοινοβουλίου το Γενάρη του 18 που μας ε, βοήθησε στην προσπάθεια μας να διατυπώσουμε το σχετικό κανονισμό. Και φαίνεται άλλωστε αυτό και στην γενική προσέγγιση του Δεκεμβρίου. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, τον εισηγητή του και όλους τους που τόσο γρήγορα ε, συνεργάστηκαν για να προχωρήσουμε σε αυτήν την αναδιαβούλευση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η έγκαιρη έγκριση της αναδιατυπωμένης οδηγίας ή ε, μάλλον του αναδιατυπωμένου κανονισμού είναι προς όφελος των παιδιών και των ε, γονέων. Γιατί ε, βοηθά να διεκπαιρεθούν πιο γρήγορα τα θέματα που άπτονται τη γονική μέρημνα. Και γι' αυτό ομόφωνα όλα τα ε, μέλη συμφώνησαν ε, το Δεκέμβριο του φακέλου αυτού. Η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου ε, του Δεκεμβρίου συγκεκριμένα αντικατοπτρίζει νομίζω και την προϋθέση του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να εκφράσουμε και την στήριξή μας προς ε, τους συζητητές, τους σκιώδεις συζητητές. Συμφωνούμε με τις αναλύσεις τους και τις σημερινές τους παρεμβάσεις και περιμένουμε και εμείς ε, να εγκριθεί τάχιστα ο κανονισμός αυτός. Αυτό είναι προτεραιότητα της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις κυρία Γκέπχαρτ και ως συγκήτριας. Σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση, θέλω να πω ότι αφορά μόνο ε, ζητήματα γονικής ευθύνης. Αυτή ήταν η πρόταση της Κομισιόν. Θέλαμε να ε, και να επιταχύνουμε τις πολύ δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες το λιγότερο κόστος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι σε θέματα αγωνικής ευθύνης καλύπτονται όλα τα παιδιά. Εφαρμόζεται ε, ανεξαρτήτως δηλαδή του καθεστώτος συμβίωση των γονέων εφαρμόζονται οι διατάξει σε όλα τα παιδιά. Για το Βρυξέλλες 2α πρέπει να δούμε πρώτα θα εγκριθεί ο αναδιατυπωμένος ε, κανονισμός για να δούμε μετά τι γίνεται με τις διατάξεις τη γονική ευθύνη, αλλά φυσικά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε συνεχώς, θα ε, παρακολουθούμε τον κανονισμό Βρυξέλλες ε, ένα και θα αξιολογούμε την ανάγκη ανάληψη ενδεχομένω δράση από την Κομισιόν. Αλλά βέβαια αυτό αφορά την επόμενη επιτροπή. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Would the council wish to take the Μήπως το Συμβούλιο να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητό ακροατήριο, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που προσεγγίζετε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης με ένα γρήγορο τρόπο και με μια ταχεία διαδικασία. Ξέρετε πως εμείς στο Συμβούλιο 7 Δεκεμβρίου καταλήξαμε στην γενική προσέγγιση. 7 Δεκεμβρίου του περασμένου έτου, και οι βασικές πτυχές αυτής της γενικής προσέγγισης είχαν να κάνουν με την κατάργηση του εκτελεστού τίτλου, με τις διατάξεις για την ε, εκτελεσιμότητα και για τις πιο ξεκάθαρες ε, κανόνες για το πώς θα εκφράζει την ε, βούλησή του το παιδί. Ε, όπως επίσης και στην κυκλοφορία των αυθεντικών ε, μέσων και συμφωνιών. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που είναι σημαντικό για τον οικογενειακό βίο είναι οι ξεκάθαροι κανόνες για την περίπτωση της παιδικής κακοποίησης στις 19 ε, Δεκεμβρίου ε, αποφασίσαμε να αναπέμψουμε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θέλουμε να προσθέσουμε όχι μόνο αυτά τα οποία είχαμε στην προηγούμενη γνωμοδότησή σας αλλά στα πλαίσια της διαφάνειας και της θεμητής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε εκ νέου τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι γιατί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες ε, Μα απομακρύνουν από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήθελε το Συμβούλιο να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρχήν να λάβει υπόψη του αυτές τις τροποποιήσεις και δεύτερον εκ νέου να γνωμοδοτήσει. Κάποιε από αυτές τι αλλαγές έχουν να κάνουν ε, την επιβολή, την αναγνώριση των αυθεντικών ε, εργαλείων, ε, μέσων με συγχωρείτε, και συμφωνιών και όπως είπαν και οι ομιλητές το κείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το Δεκέμβριο το, Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο ε, δίνει προστιθέμενη αξία έτσι ώστε να έχουμε επιταχυμένες διαδικασίες σε θέματα αγωνικής επιμέλειας και ευθύνη. Εδώ θα μπορούσα να ευθυγραμμιστώ με τα όσα είπε ο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η αναπομπή είχε να κάνει μόνο με τι πτυχέ αυτή τη γονική φροντίδα και η δική μας άποψη στο Συμβούλιο είναι πως το κείμενο όσο έχει σήμερα στη γενική προσέγγιση δίνει προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, το συμφέρον του παιδιού είναι μια αρχή την οποία ακολουθούμε ε, καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κανόνων για την ακρόαση του παιδιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όπως είπε και ο εισηγητής, η γενική προσέγγιση Συμβουλίου έλαβε υπόψη σημαντικές ιδέες και αρχές που ήταν παρούσες ε, στην γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ήταν η, η, η, η ακρόαση του παιδιού και ε, τα θέματα που άπτονται της ε, διασυνοριακής και και πιστεύουμε πως και εσείς και εμείς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε τον ίδιο στόχο. Δεδομένη σημασία αυτής της ε, νομοθεσίας για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για όλες τις οικογένειες, θεωρούμε πως αποτελεί υψηλής προτεραιότητας ε, φάκελο για το Συμβούλιο και τη Ρουμανική Προεδρία και πραγματικά εκτιμάμε ιδιαίτερα την ταχύτητα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σκοπό να ανταποκριθεί στη διαδικασία και περιμένουμε τη νέα γνωμοδότησή σας για το, κοινό, για το νέο αυτό κείμενο το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη, επαναλαμβάνω, την επίγουσα φύση του φακέλου και τη σημασία που έχει για Στόχο και τα παιδιά. Στόχος του Συμβουλίου είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο του 2019 και στα πλαίσια αυτά καλό θα ήταν να έχουμε την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ε, μέσα στι προθεσμίε. Πιστεύω πως ο Σκιώδης αντιμετώπισε και αυτό κάποια από τα ζητήματα και εδώ πρέπει να ευθυγραμμιστώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, thank you as well. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ξέρετε κι εσείς πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει νέο συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού. Είναι η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, η οποία μόλις μπήκε στην αίθουσα. Οπότε καταρχήν θα ήθελα να τη συγχαρώ για το διορισμό της και θα ήθελα να σας δώσω και το λόγο για 60 περίπου δευτερόλεπτα γιατί περνάμε τώρα πολύ σύντομα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ. Ε, λυπούμε πάρει αλλά ψήφιζα σε μια άλλη επιτροπή. Θα είμαι πολύ σύντομη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Αυστριακή Προεδρία κατάφερε να καταλήξει συμφωνία για τον κανονισμό. Πολλούς φίλους βλέπω εδώ. Τι ωραία. Χαίρομαι που σας βλέπω. Χαίρομαι που επιτεύχθη συμφωνία και με βέβαιο ότι στα ικανά χέρια του Αντέου ε, με την επιτυχημένη αυτή διαδικασία θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε και ελπίζω να γίνει αυτό πράξη μέχρι το τέλος της τα σχετικά ως συντονίστρια για τον των παιδιών θεωρώ ότι είναι θετικό που έλειψαν υπόψη και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις διασυνοριακές αρπαγές, τις διεθνείς αρπαγές παιδιών που πλήττουν την καθημερινή ζωή των ε, ε, παιδιών φυσικά ε, και των οικογενειών τους, αλλά κυρίως είναι τραυματικές εμπειρίες για τα παιδιά. Λίγα πράγματα μόνο. Να πω ότι είναι πολύ θετικές προσπάθειες που έγιναν για τις διαδικασίες αν έχουμε μία αρπαγή παιδιού διευκρινήσεις για τη διάρκεια της δικασίας, ε, τις διορίες, ε, τα, ε, τις προσφυγές. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό θέμα είναι η υποχρέωση το δικαστήριο να το παιδί. Δηλαδή, φωνή του παιδιού μπορεί να ακουστεί. Αυτό είναι θετικό. Και το τελευταίο σημείο βέβαια είναι σημαντικό κατ' εμέ το ότι αυτός ο κανονισμός ενθαρρύνει, παροτρύνει τη διαμεσολάβηση, τη διαιτησία, τις διαβουλεύσεις και την αλλακτική επίλυση της διαφοράς. Σε ό,τι διαφορά την ε, διαμεσολάβηση νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένας ο πόρος να προτείνει βέλτιστες πρακτικές, να βοηθήσει τα παιδιά. ώστε να επιληφθούν με καλύτερο τρόπο οι σχετικές διαφορές. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Ταντέους. Ευχαριστώ που ήρθες και για τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ δεν φαίνεται να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό το σημείο και βεβαίως ε, θα προχωρήσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ βάλτε την κάρτα σας στο ειδικό μηχάνημα. Η Κυρία Ρεντέν, ναι, ε, έρχεται τώρα ο σύμβουλός μας με, την, με το κατάλογο ψηφοφοριών. Αν μπορούμε να περιμένουμε δύο λεπτά, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Ε, ε, You can follow the EPP if you wish, you know. So... Μπορείτε να ακολουθήσετε το ΕΛΚ αν το επιθυμείτε. So we have all the voting this except Λοιπόν, έχουμε όλους τους καταλόγους εκτός από το SPC. Εάν δούμε το SPC τελευταίο, μπορούμε να ξεκινήσουμε. So Let's uh, let us begin item number seven. Λοιπόν, ξεκινούμε με το σημείο 7. Κανόνες για την ε, άσκηση των δικαιωμάτων copyright και σχετικών δικαιωμάτων. Ο κ. Λεμπρετών είναι ο εισηγητής. κ. Λεμπρετών, θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Όχι, Πρόεδρε, νομίζω δεν χρειάζεται. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που προτάθηκαν από την νομική υπηρεσία. Πολύ ωραία. Θα είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία.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 μέλη του ΕΛΚ εδώ. Αν θέλετε μπορώ να μην ψηφίσω εγώ. Είμαι ρυθμένο να μην ψηφίσω. Εντάξει. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας Μάλιστα, εγκρίνεται λοιπόν. Πάμε τώρα στο σημείο 8. Μια προφορή, προσωρινή συμφωνία να σας πω ότι ο έκτος και τελευταίος τρίλογος έλαβε χώρα στις 13 Δεκεμβρίου και στον τρίλογο αυτό τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μετά τον πέμπτο τρίλογο και το πεδίο της, ε, της επέκτασης της, ε, της έννοιας της χώρας προέλευσης. Ε, υπήρξε συμφωνία και για τα διάφορα πολιτικά εκκρεμή ζητήματα, την μεταβατική περίοδο, την ημερομηνία μεταφοράς και την τρίτη αναθεώρησης. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Uh, please, please, so, sorry, listen to me. We... Ναι, ακούστε με λίγο. Θα ξεκινήσουμε εκ νέου την πληροφορία για να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούν τα διάφορα μηχανήματα. Ναι, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς ψηφίζουμε, γιατί εγώ μόλις μπήκα στην αίθουσα. Ε, ε, ποιος είναι ο εισηγητής, ποια είναι η γνωμοδότηση. Ε, επακριβώς. Euh, Μόλις έφτασα. Ναι, είναι η προσωρινή συμφωνία μετά από τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για το ΣΑΠΚΑΠ. Δεν ακούω. Σας It's item 8. Okay, thank you. Εντάξει, ευχαριστώ. Yes, we, we restarted the vote. Λοιπόν, ξεκινάει εκ νέου ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Yes. And that has been adopted. Εγκρίνεται λοιπόν και προχωράμε στο σημείο 9 ψηφίζουμε για το πρωτόκολλο υπαριθμών 3 εδώ προσωρινή συμφωνία μετά από διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ο κύριος Βέλκεν θέλει να, να, κάνει κάποια εισαγωγή για αυτόν τον ε, τετράλογο που έλαβε χώρα. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Close it. And that has been adopted. Uh, then... Εγκρίνεται και προχωρούμε στο 10. Έκθεση της κυρίας Νίμπλερ. Και εδώ ψηφίζουμε επί μιας προσωρινής συμφωνίας. Κυρία Νίμπλερ, θέλετε να πείτε κάτι? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω θερμό όλους τους κοιόδες για την πολύ καλή συνεργασία. Συναντηθήκαμε ανεπίσημα πολλές φορές ε, και διαμορφώσαμε εδώ την θέση μας. Ε, πολύ καλά προχώρησε και το μέρος διάλογος ευχαριστώ όλους τους και ηγητές για την τεράστια και πολύ σημαντική συνεισφορά ώστε ε, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες και δι' τους νέους ε, να έχουν ε, μια καλύτερη ευκαιρία και να είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες οικονομικές τους δυσκολίες. Ξέχασα να συγχαρώ τον κύριο Βέλκεν προηγουμένως, το συγχαίρω τώρα να ψηφίσουμε λοιπόν εκ νέου ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. So that has Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Νίμπλερ. Και περνάμε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 μετά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 όχι δεν ψηφίζουμε το 17 ε, επί της 17 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ για την τροπολογία 80 ψηφίζουμε εγκρίνεται 81 υπέρ συγγνώμη δικό μου το λάθος 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 όχι καταπίπτει 82 όχι α όχι δικό μου λάθος πάλι ψηφίζουμε επί της 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ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 κατά. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 89, ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε για την 96 παρακαλώ ψηφίζουμε απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκατό υπέρ κατά αποχές εδώ πρέπει να το δούμε αυτό να το παληθεύσουμε εκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 102. εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά να ρωτήσω παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι 4 υπέρ. Μπορεί να ψηφίσει το ΕΛΚ. Μπορεί να ψηφίζει δηλαδή και η δεύτερη σειρά, αν γίνεται, του ΕΛΚ. ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ε, δεν μπορεί να... θέλω να διακόπτω την α, ψηφοφορία, αλλά θέλω να ξέρω από τον κόσμο να ψηφίσει. Είναι θέμα πειθαρχίας. Ναι, τώρα να διακόπτετε εσεί και να σου λέτε ψηφίστε, μην ψηφίζετε, ψηφίζετε. Κάνετε επαλήθευση ηλεκτρονικά, εάν θέλετε. Τώρα να μας λέτε να ψηφίζετε νομίζω ότι είναι περιβολικό. Ναι, ευχαριστώ που κάνετε τη δουλειά μου, κύριε Πίντο. Είμαστε σε 104, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 23, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά 112 επαλήθευση. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Ωραία. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 113. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά Ας ε, επαληθεύσουμε την 116. Ψηφίστε παρακαλώ. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 119 παρακαλώ εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία 120 υπέρ κατά Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 120. Εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει αυτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ το 44 πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη 48 παρακαλώ ψηφίζουμε εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά να ελέγξουμε και την 50 παρακαλώ απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ ναι, 56 υπέρ κατά Να ελέγξουμε και την 57 λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ Κατά. Να ελέγξουμε τη 12 παρακαλώ. Μάλιστα. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί του συνόλου της γνωμοδότησης. Απορρίφθηκε. Οπότε φαντάζομαι δεν μπορώ να δώσω χατέρα στον κύριο Λεμπρετών. πράσινοι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν τώρα για το επόμενο θέμα. Πολύ ωραία. So we vote on the report of Mr. De Grandes. Ψηφίζουμε για την έκθεση του κύριου De Grandes Pascual. Τα επιπλέον πιστοποιητικά προστασία για τα ε, ιατρικά προϊόντα. Ε, Δεν ξέρω αν ο εισηγητής θέλει να λάβει το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ξέρετε πως ο φάκελος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εδώ αντιμετωπίσαμε δύο ε, οι κατηγορίες συμφερόντων που όλα χρησιμοποιούνται και βεβαίως όλες οι ομάδες προσπαθήσαμε να δείξουμε ευελιξία, να δεχτούμε ε, το κομμάτι που έχουν δίκιο πάντα οι αντίπαλοι μας, να συμβιβαστούμε και ελπίζω πως το αποτέλεσμα είναι υπέρ της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμβιβαστική 1 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται We go to 196. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. NV25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2.14 υπέρ 240, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά. Το 240 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική και οκτώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική εννέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ. Κατά αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονικά και τη συμβιβαστική α. Παρακαλώ. Εγκρίνεται. Yes. Compromise 10. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην 27, τροπολογία 27, υπέρ, κατά. Αποχές. Παρακαλώ την 27, θα ήθελα να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. False. NV2. Λοιπόν, NV2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα έλεγα απορρίπτεται, αλλά επειδή είδα τόσο λίγα χέρια, θέλω ηλεκτρονικά να κοιτάξουμε πάλι την NV2 εγκρίνεται. Είναι τα ένα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ την 32 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. «33 και 34 υπέρ». Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ 33 και 34 μαζί. 33 και 34. Απορρίπτεται. NV3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ίντα 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν την ίντα 3 ηλεκτρονικά παρακαλώ ίντα 3 ηλεκτρονικά εγκρίνεται συγχωρέστε με 35 υπέρ κατά Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 35. Απορρίφθηκε. Είναι τα 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, παρακαλώ πολύ ηλεκτρονικά και την τα 4. Sorry, my mistake. Εγκρίνεται. 36 in favor. 36 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά Μπορώ να δούμε, μπορούμε να δούμε ηλεκτρονικά την 137 παρακαλώ Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, λέω. Αλλά καλύτερα να το δούμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι. Τη συμβιβαστική Β, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται λοιπόν. Πάμε τώρα λοιπόν στην 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV19 υπέρ κατά. Παρακαλώ τη 19 να τη δούμε μαζί. Uh, that Compromise 24. In... 24 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 146. Δεύτερο τμήμα. Εκατόν δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Θα Θα ήθελα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν. Για το σύνολο του σχεδίου άρχεται η ψηφοφορία. Uh, I Πέρας. Εκκρίνεται. Θα ήθελα να συγχαρώ λοιπόν αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε και την απόφαση των δύο οργανικών ε, διαπραγματεύσεων στις οποίες θα μπούμε τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κύριε Τεγκράντες Πασκουάλ. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με την έκθεση της κυρίας Ρόζιερ για το σχέδιο δράσης και την προσχώρηση στην πράξη της Γενέβης για τις ονομοσίες προέλευσης και τους γεωγραφικούς προ... διορισμούς. Τροπολογία 30 υπέρ. Against. Κατά. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Συγγνώμη. Θα επαναλάβω την ψηφοφορία από την αρχή. Λοιπόν, τροπολογία 30. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Είναι τα πέντε ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ένα ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική δύο ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία για 16 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα 12 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολή 48. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τα 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολή 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Ποιες εγκρίνεται. Είναι τα 1. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε την 20 παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Συμβαστική αναψήφη υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, δεν έπρεπε. Πρέπει να την είχα θέσει ψηφοφορία. Τέλο πάντων. Συμβαστική 2. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ εγκρίνεται 7 ψηφιπέ κατά εποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σχέδιο της έκθεσης τώρα συνολικά ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίθηκε απόφαση ανάξης διαπραγματεύσεων διοργανικών διαβουλεύσεων ηλεκτρονικά. Κύριε Υπάρχει ένα λάθος στον κατάλογο τη ψηφοφορία. Δεν καλυπτώ όταν από τη συμβαστική 4 ή 8 η τροπολογία 8 και έπρεπε να έχει τεθεί σε ψηφοφορία, πιστεύω. Πρόεδρος. Ναι, άρα έχει λάθος η, η λίστα ψηφοφορίας. Άρα να επανέλθουμε στην τροπολογία 8, το συγγνώμη, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε και τώρα Ψηφίζουμε την εντολή έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ηλεκτρονικά. Εγκρίθηκε συγχαρητήρια στην κυρία Ροζιέλ. Και τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση του Καβαντά. Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Όλαφ. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1361, ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνονται. 62, ψήφι υπέρ, κατά, όχι, 62, 62, ψήφι υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 63, υπέρ, κατά να ελέγξουμε την 63. Ε, yes. Slightly Με μικρή διαφορά εγκρίνεται. 65 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 ψήφι περ. 66. Τι θέλετε, να ελέγξουμε την 65. Ναι, ας το κάνουμε. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. 66 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 ψηφίπερ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 14 και 69 ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνονται. 70 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 70. εγκρίθηκε 71 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 72 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 73 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 74 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 75 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 76 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 82 ψήφι ΠΕΡ κατά εποχές θα έλεγα καλύτερα να ελέγξουμε πράγματι απορρίπτεται 84 ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές απορρίπτεται 85 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 και μάλλον 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 ψηφιπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 28 ψηφιπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 29 ψηφιπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 30 ψηφιπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται 32 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 ψήφι περ. κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 ψήφι περ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 ψήφι περ. κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 9 ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Τροπέ 40 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 43 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά Εποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται το σχέδιο της γνωμοδότησης ε, ονομαστικά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Καβαντά. Καλώς ήρθατε κιόλας. We continue by the report of Madame Bergeron. Έκθεση Bergeron. Συνεργασία μεταξύ Γιώργης και Γεωργίας, ηλεκτρονική και μία ψηφοφορία άρχεται.